με τις ψηφοφορίες. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε την έκθεση του κύριου Μορέιρα. Την συμπερίληψη δηλαδή της ε, Γρυλανδίας ε, στο σύστημα ε, πιστοποίησης Κίμπερλι. Θα γίνει ονομαστική η ψηφοφορία και άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, ερωτώ. Ψηφίσατε όλοι λοιπόν. Θα αναμείνω μερικά δευτερόλεπτα. Και έτσι τώρα πέρας ψηφοφορίας πλέον. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Και τώρα στη συνέχεια περνάμε στην δεύτερη έκθεση στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται πάλι για μια έκθεση του κυρίου Μορέιρα, αυτή τη φορά για την συμμετοχή της ε, Γρυλανδίας στο σύστημα πιστοποίησης διαδικασίας Κίμπερλι. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Η έκθεση εγκρίθηκε. Η επόμενη έκθεση είναι η έκθεση της κυρίας Sharon Bowles. Μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την, Ευρω... την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. η έκθεση. Επόμενη έκθεση είναι η έκθεση του κ. Βέρνερ Κούν για τη συμφωνία του Cape Town της πόλης του Ακροτηρίου 2012 για την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλου του Τόρε Μολίνος ε, του 1993. Η Διεθνή Συμφωνία όσον αφορά τη Συμφωνία 1977 υπέρ παρακαλώ κατά, κατά αποχές Κατά, παρακαλώ. Μια τεχνική παρατήρηση από σας παρακαλώ. Το να αλλάζουν οι θέσεις και να μην ενημερώνονται οι ευρωβουλευτές. Έχω ένα άτομο που κάθεται εκεί που έπρεπε να ψηφίζω. Δεν ψήφισα και από την αρχή γιατί δεν μπόρεσα να καθίσω στο έδρανό μου. Και παρακαλώ τουλάχιστον να αναγγέλλεται αυτό στους ευρωβουλευτές όταν υπάρχει αλλαγή θέσεως. Θα ήθελα να ξέρω πού κάθομαι τώρα. Ε, Κυρίες και κύριοι, και για την θέση στην οποία κάθεται ένας ευρωβουλευτής ε, και που μπορεί να ψηφίζει όμως και σε από άλλο έδρανο. Δεν πρέπει υποχρεωτικά να ψηφίζει από την αρχική θέση του. Έκθεση λοιπόν του κυρίου Βέρνερ Κούν που εγκρίθηκε. Στη συνέχεια έχουμε την επόμενη έκθεση της κυρίας Εύα Λίχτενμπεργκ. 29η ετήσια έκθεση όσον αφορά τον έλεγχο εφαρμογής δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Η έκθεση εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε. Επόμενη έκθεση. Έκθεση Bernhard Ραπκάι. Έτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας ε, της Λάρα Κόμη. Λάρα Κόμη. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές η έκθεση εγκρίθηκε επόμενη έκθεση έκθεση σε Βίξτροεμ Έτηση αίτηση άσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Σμπίγνιεφ Ζόμπρο σύμφωνα με την το 175 έχει τον λόγο κύριο Ζόμπρο Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, να σας ζητήσω να αρθεί η κοινοβουλευτική μου ασυλία. Είμαι κατά της βουλευτικής μου ασυλίας. Ζητώ να αρθεί εξ ονόματός μου η κοινοβουλευτική μου ασυλία. Και αναμένω ότι θα ακολουθήσετε το έτοιμά μου. Ευχαριστώ. Okay. Εντάξει, πολύ καλά. Έχετε τον λόγο εσείς παρακαλώ. Διαδικαστικό κύριε Πρόεδρε γιατί αναφέρεται και το όνομά μου στην ε, έκθεση για την άρση της κυρίας ε, Κόμη. Ε, ε χαίρομαι, δόθη ο λόγος στον προλαλήσαντα, ενώ εμένα μου το αρνήθηκαν. ο κύριος Ραπκάη και η πλειοψηφία της Επιτροπής θεωρεί ότι στην περίπτωση της κυρίας Κόμη όταν μιλάει για οικονομία φέρεται ως Ευρωπαία Βουλευτής, ενώ όταν εγώ μιλάω για την μετανάστευση, ε, ύψιστο θέμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν είμαι Ευρωπαίος Βουλευτής. Δύο μέτρα και δύο σταθμά επομένως. Δεν θα ανοίξουμε συζήτηση τώρα εκ νέου επ' αυτού για μια έκθεση που ήδη έχει εξεταστεί. Όμως θα καταχωρηθεί στα πρακτικά οπωσδήποτε η παρατήρησή σας. ο κύριος Ζόμπρο έδωσε κάποιες διευκρινήσεις τώρα σε σχέση με το αίτημα το οποίο διατύπωσε. Τώρα θα ψηφίσουμε την έκθεση Βίξτραμ υπέρ. Ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές. Η έκθεση αυτή εγκρίθηκε. Και συνεχίζουμε με την επόμενη έκθεση του κυρίου Μπέρναρντ Ραπκάη. Πρόθεση της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα θα ψηφίσουμε για τις ε, τροπολογίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Υπέρ παρακαλώ αυτόν. Κατά. Αποχές. Η έκθεση εγκρίθηκε λοιπόν. Οι τροπολογίες, ε, συγγνώμη, εγκρίθηκαν τώρα. Η τροπολογία 16. Υπέρ κατά αποχές η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε ακολουθεί η τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η τροπολογία στην συνέχεια η τροπολογία 2 και 11 της Κοινοβουλικής Επιτροπής υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. Τώρα ονομαστική ψηφοφορία. Μάλιστα. Θα ελέγξουμε όπως ζητήσατε. Ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκαν οι τροπολογίες. Τροπολογία 51-52 καταπίπτουν αυτές τις τροπολογίες. Ψηφίζουμε για την 48 και 49 τώρα, υπέρ αυτών. Κατά αποχές εγκρίθηκαν. Τώρα η τροπολογία της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν οι τροπολογίες αυτές. Και τώρα ονομαστική ψηφοφορία ακολουθεί με ονομαστική κλίση για το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Και έχουμε τώρα και την έκθεση της κυρίας Σαγιά που ακολουθεί. Ταξινόμηση και επισήμανση συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τώρα θα ψηφίσουμε για την ομάδα υπαριθμό 2, κατηγορία 2, τροπολογίες 1 και 19. Όχι, ο πρόεδρος διορθώνει, καταπίπτει αυτό. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε την πρόταση της Επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Και τώρα θα ψηφίσουμε την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Και θα ψηφίσουμε τώρα την έκθεση Γκαλό. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα και χορήγηση αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχύω για μουσικά έργα και επιγραμμικές χρήσεις. Τροπολογία 170. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ακολουθεί η τροπολογία της Επιτροπής ε, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και ακολουθεί τώρα η πρόταση νομοθετικού περιεχομένου ψηφίσματος, ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Και περνάμε στην έκθεση Μακάθη. Ποινικέ κυρώσει για καταχρήσει εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγηση αγοράς. Ψηφίζουμε την τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τώρα την πρόταση της Επιτροπής ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τώρα ψηφίζουμε την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Πρόταση ψηφίσματος ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε το νομοθετικό ψήφισμα. Και τώρα θα ψηφίσουμε την έκθεση Βάλεαν, επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακές υποδομές. Ψηφίζουμε την τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 39 ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ πέρας της ψηφοφορίας η τροπολογία αυτή απερίφθη και τώρα στη συνέχεια τροπολογία 40. Ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Η τροπολογία αυτή απορρίφθηκε. Και στη συνέχεια έχουμε την τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τώρα η τροπολογία 41 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε η τροπολογία αυτή. Και ψηφίζουμε τώρα η τροπολογία 42. Ονομαστικά πάλι άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. η τροπολογία αυτή απορρίφθηκε. Τροπολογία 43, ονομαστικά πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε η τροπολογία αυτή. Και ακολουθεί τώρα η ψήφιση της πρότασης Επιτροπής. Ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε η πρόταση. Και θα ψηφίσουμε τώρα την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου <clears throat> ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε η νομοθετική πρόταση ψηφίσματος. Και περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Αγιάλα Σέντερ από πλευρά του ελεγκτικού συνέδριου σε σχέση με το ελεγκτικό συνέδριο. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1 υπέρ. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Προεδρεύων. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στην έκθεση Αγιάλα Σέντερ και πάλι πρόκειται για τον ορισμό μέλους στο ελεγκτικό συνέδριο, τον ορισμό του κυρίου Κλάους Χάινερ Λένε στο ελεγκτικό συνέδριο. Θα ψηφίσουμε λοιπόν σε σχέση με αυτό το αίτημα με μυστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας. και αποτέλεσμα. Ο κύριος Λένε επικυρώθηκε στη θέση αυτή ως μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, ε, εγκρίθηκε ο ορισμός του και έτσι τοποθετείται στο ελεγκτικό συνέδριο. Επιτρέψτε μου <clears throat> κύριε Λένε και εξ μου να εκφράσω θερμά συγχαρητήρια προς εμάς. Κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό επανερχόμεθα στην έκθεση της κυρίας Αγιάλα Σέντερ που αφορά το ελεγκτικό συνέδριο. Και τώρα ζητώ από την κυρία Γιάλα Σέντερ για δύο λεπτά να μας εξηγήσει τα σχετικά παρακαλώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Απλά και μόνο ήθελα και δεν υπήρχε αυτή η ευκαιρία να γίνει σύντομα μια συζήτηση για κάτι το οποίο θα μπορούσε να ενδιαφέρει όλους. Απλά θέλω να ευχαριστήσω όλους για το έργο που επιτέλεσαν σε σχέση με αυτή την έκθεση και ιδιαίτερα επίσης τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου που στο πρόσωπο του κυρίου Καλτέρα το επικεντρώνω αυτό το έργο που έγιναν σημαντικές μεταρρυθμίσεις ώστε το ελεκτικό συνέδριο να γίνει ένα πιο εξειδικευμένο και πιο αποτελεσματικό έργανο, όργανο το ελεκτικό συνέδριο που θα ανταποκρίνεται κυριότερα στα αιτήματα των κυριότερων πελατών του που είμαστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο αλλά επίσης να υπάρχουν και στοιχεία εμπιστοσύνη προς τους πολίτες ότι τουλάχιστον κάποιο επιτηρεί για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Έγινε αυτή η έκθεση και θελήσαμε να προχωρήσουμε πιο πέρα και να προκαλέσουμε ώστε να υπάρξουν δημιουργικά στοιχεία, ώστε να υπάρξει προσπάθεια να επιληθεί το πρόβλημα σε σχέση με την αρνητική πιστοποίηση, σε σχέση με την βελτίωση πραγμάτων όσον αφορά την, το ελεγκτικό συνέδριο, ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο πιο κοντά στα μελήματα για την ευρωπαϊκή πολιτική. Και έχουν βελτιωθεί νομίζω αυτά τα πράγματα. Και επίσης είναι απόδειξη ο, ο ορισμός του κυρίου Λένε σήμερα στο ελεγκτικό συνέδριο. Ε, βελτίωση και των κριτηρίων για την επιλογή υποψηφίων. Ζητώ λοιπόν να υποστηριχθεί τροπολογία 1, όπου ζητείται η βελτίωση. Αυτό που από πλευρά Κοινοβουλευτική Επιτροπή κάναμε, ζητώ συγγνώμη και ζητώ συγγνώμη για την παρέμβασή μου αυτή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέμβασή σα και τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε για την τροπολογία 1. Είναι μια εναλλακτική τροπολογία υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε η τροπολογία. Μάλιστα. Μπορούμε και να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά επ' αυτής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Και ως εκ τούτου στη συνέχεια θα ψηφίσουμε το ψήφισμα της Επιτροπής, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στο σύνολό, σύνολό του υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε η πρόταση. Και στη συνέχεια περνάμε στην έκθεση του κυρίου Κάριμ. Βελτίωση τη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την επικουρικότητα και αναλογικότητα σε σχέση με την καταλληλότητα κανονιστικού πλαισίου. Τροπολογία 1. Ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε η τροπολογία αυτή. Ψηφίζουμε την τροπολογία 2, ονομαστικά πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε η τροπολογία αυτή. Τώρα η τροπολογία 3, ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Η τροπολογία αυτή απορρίφθηκε. Ακολουθεί η τροπολογία 8, δέλτα, ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Η τροπολογία αυτή απορρίφθηκε. Και ακολουθεί η τροπολογία 9, ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε η τροπολογία. Τροπολογία 4. Ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Η τροπολογία απορρίφθηκε. Και τώρα έχουμε την τροπολογία 5 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Η τροπολογία απορρίφθηκε. Ακολουθεί η τροπολογία 6 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε η τροπολογία. Ακολουθεί η τροπολογία 10. Δέλτα. Ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Η τροπολογία αυτή απορρίφθηκε. Και στη συνέχεια περνάμε στο εδάφιο 36 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε το πρώτο τμήμα. Ακολουθεί το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε το δεύτερο τμήμα. Τώρα η τροπολογία 7 ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Η τροπολογία εγκρίθηκε. Και θα ψηφίσουμε τώρα την πρόταση ψηφίσματος στο σύνολο της ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε η πρόταση. Κυρίες και κύριοι, θα ακολουθήσει τώρα η επίσκεψη του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 12.30 λοιπόν. Ευχαριστώ. Okay. Thank you.